Hello everyone and good evening. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι. Ελπίζω να μην μας γίνει συνήθεια στο Στρασβούργο κάθε Δευτέρα βράδυ, αλλά πάση περιπτώσει δεν εξαρτάται από εμά. Είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ημερήσια διάταξη. Αντιρρήσεις. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Έχουμε κάποια επίγοντα ζητήματα, ψηφοφορίες για παράδειγμα. Και γι' αυτό έκτακτη συνεδρίαση θα έχουμε στις 25 Οκτωβρίου, που είναι πέμπτη στο Στρασβούργο, από τις 8.30 το πρωί και λυπάμαι για το πρωινό της ώρας. Πέμπτη απόγευμα 18 Οκτωβρίου τώρα δεν θα έχουμε συνεδρίαση. Το πρωί, ναι. Το σχέδιο μερίσιας διάταξης θα μοιραστεί έγκαιρα. Έχετε επίσης την έκθεση για την αποστολή μας που επισκέφτηκε τις Γαλλικές Άλπεις πρόσφατα, Σαβουά και Ιζέρ, αυτές τις δύο περιφέρειες, όσον αφορά την παρουσία λύκων. 12 και 13 Ιουλίου ήταν αυτή η αποστολή. Σήμερα έχουμε 20 γλώσσες, να ξέρετε, διερμηνία και ευχαριστεί τους διερμηνείς η Πρόεδρος. Η ηλεκτρονικά έχετε τον φάκελο με όλα τα έγγραφα και μεταδίδεται στο διαδίκτυο επίσης η συνεδρίασή μας. Έχετε επίσης και τα πρακτικά μας στις 20 και 21 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και τώρα, όσον αφορά τις ε, διαοργανικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Για το θέμα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ο πρώτος ε, τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα πιο πολιτικά ζητήματα που διακυδεύονται στην υπόθεση αυτή. Και παρά τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλή ατμόσφαιρα και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Για το αντίστοιχο θέμα για το πουλ, αποφασίσαμε να συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο η συζήτηση για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό που θα πάει στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα γίνει 8 Οκτωβρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Ελπίζω να έχουμε καλύτερα νέα τότε, γιατί προς το παρόν το Συμβούλιο φαίνεται να είναι πολύ ξεροκέφαλο και να μην θέλει να μετακινηθεί από τη θέση του όσον αφορά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο νομοθετικό ζήτημα που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, που είναι το πρόγραμμα Invest EU, με εισηγητή τον κύριο Μπέλετ που είναι μαζί μας. Έχετε το λόγο κύριε Μπέλετ, παρακαλώ. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, έτσι, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το Invest EU είναι ο διάδοχος του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού δηλαδή Προγράμματος Στρατηγικών Επενδύσεων. Η δικιά μας η Επιτροπή συνεισφέρει, παρόλο που οι αρμόδιες επί της επιτροπές είναι η Προϋπολογισμών και η Οικονομική Επιτροπή. Εμείς γνωμοδοτούμε και η Ρέτζι και η Καλτ πολιτισμού. Θέλω λοιπόν από αυτής εξ αρχής ότι στο σχέδιο αυτό κειμένο μου θέλουν να επικεντρωθώ στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα με διάφορα προγράμματα τα οποία λειτουργούν εκ Για παράδειγμα, στο παράρτημα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ένα παράδειγμα που είναι η κεφαλαιακή διευκόλυνση. Και το άλλο είναι οι ιδιωτικέ επενδύσεις για τον μηχανισμό ενεργειακής απόδοσης. Υπάρχει και το κόσμο. Θέλω να πω υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά ε, μέσα, μηχανισμοί και στόχος μας είναι όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε σε ένα πρόγραμμα. Ο στόχος λοιπόν είναι πολύ καλός και φυσικά και τον στηρίζουμε. Είναι μια μεγάλη όμως μεταρρύθμιση αυτή. Τα κύρια στοιχεία της πρότασης αυτής είναι το Ταμείο Invest EU που αποτελεί εγγύηση για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά παράθυρα, δηλαδή τέσσερις διαφορετικοί τομείς πολιτικής μέχρι 11 εκατομμύρια. Υπάρχει η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφοποίηση, 11 δισεκατομμύρια βιώσιμη υποδομή, 11 δισεκατομμύρια μικρές και μισές επιχειρήσεις, 11 δισεκατομμύρια και τέλος κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες, 4 δισεκατομμύρια. Όπως είπαμε ήδη, για την διαχείριση στα πλαίσια του ΕΦΣΙ, την διαχείριση των εγγύσεων την είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στα πλαίσια του Invest EU, τη διακυβέρνηση του προγράμματος προβλέπεται να γίνει και με άλλες ε, τράπεζες. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά λοιπόν. Δεν θα είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το είπαμε και στην αρχή εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ αποκλειστικά στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της δικιάς μας Επιτροπής. Και τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση του Ταμείου τα αφήνουμε στους συναδέρφους στην Επιτροπή Ευρωπολογισμών και στην Οικονομική Επιτροπή. Παρ' όλο αυτό όμως πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την διαδικασία για να ξέρουμε πώς θα έχει αυτή η διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ παρούσα, οπότε θα θέλαμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην διαδικασία της διακυβέρνησης. Τώρα, σε τρία θέματα θέλω να επικεντρωθώ, και που ενδιαφέρουν πολύ εμά. Το ένα είναι η βιωσιμότητα. Μέσω του επενδυτικού αυτού ταμείου, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το δυοσημότητα. Δεύτερον, να ε, λαμβάνεται υπόψη διάσταση του κλίματος ε, σε όλες τις πολιτικές, όλες τις αποφάσεις και το τρίτο βέβαια είναι η κλιματική αλλαγή. Εμείς ε, καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα. Το θέλουμε αυτό, αλλά θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει συγκεκριμένες απαιτήσει για όλα τα παράθυρα, όχι μόνο για τις υποδομές. Για όλους τους τομείς πολιτικής λοιπόν. Και όχι μόνο ε, εκεί που το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι σε ένα από τα τέσσερα παράθυρα. Θέλουμε ελάχιστες προδιαγραφές βιωσιμότητες για όλους τους τομείς πολιτικής, για όλα τα προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται από το Invest EU. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για μένα. Και το τονίζω στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησής μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να το πω και αυτό κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, προβλέπει με την πρότασή της κάποια εξαίρεση για μικρά προγράμματα, τα οποία θα καθοριστούν βάσει καταξουσιδότηση πράξεων. Θέλουμε να τις διατηρήσουμε αυτές τις εξαιρέσεις. Τώρα είπαμε για τη βιωσιμότητα, το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η διάσταση του κλίματος. Πώς θα σωματώνει τη διάσταση του κλίματος σε όλες τις πολιτικές. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν λέω τίποτα καινούριο, και να συμμορφωθούμε με τη γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήδη εγκρίθηκε το Μάιο που μας πέρασε, με ψήφισμα της 30 η Μαΐου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εκεί ήδη αποφασίσαμε να έχουμε δαπάνες πιο φιλόδοξες όσον αφορά το κλίμα και προτείνουμε 35% να καθοριστεί δηλαδή ένα στόχος 35% για το πρόγραμμα InvestEU. Επιπλέον από αυτόν τον φιλόδοξο στόχο θέλουμε επίσης να έχουμε και μια αξιόπιστη και διαφανή μέθοδο παρακολούθησης της διαδικασίας. Μας απασχολεί κάπως το γεγονός ότι στα προγράμματα που έχουμε τώρα, στο τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μερικές φορές δεν έχουμε ούτε καν 20% δαπάνες για το περιβάλλον, για το κλίμα. Και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του Ιουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο στόχος δηλαδή του 20% δεν επιτυχάνεται καν. Τώρα λοιπόν θέλουμε να βάλουμε ως νέο στόχο το 35% αλλά να υπάρχει και μία αξιόπιστη μέθοδος παρακολούθησης για να βλέπουμε κατά πόσο επιτυχάνεται αυτό το 35% ή όχι. Και σε αυτό να προσθέσω ότι έχω, επενδύσει και, έχω συγγνώμη, υποβάλει και μία τροπολογία με την οποία ξεκαθαρίζω ότι όσον αφορά αυτήν την αξιόπιστη μέθοδο παρακολούθησης θέλουμε κάτι ξεχωριστό για το κλίμα και κάτι ξεχωριστό για τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Να ξέρουμε δηλαδή να έχουμε μια μέθοδο παρακολούθησης αξιόπιστη για το τι δαπανάτε για το κλίμα και τι για τους υπόλοιπου στόχου που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Αναφέρθηκα λοιπόν στη βιωσιμότητα, αναφέρθηκα στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω εδώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, είναι ότι οι επενδύσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας ε, φυσικά και αυξάνονται. Όμως υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας όσον αφορά την παραγωγή με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Και θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε ε, τα προγράμματα τέτοιων επιχειρήσεων που παράγουν με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Και ιδιαίτερα προγράμματα που είναι μεν χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά που ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος για αυτές. Οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και να υπάρχουν πληροφορίε σχετικά με την αποφυγή του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει ε, βιομηχανικά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνει την πρόσβασή του σε χρηματοδοτική στήριξη. στα πλαίσια των διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε επίσης να βιαστούμε. Κάνουμε μια έκκληση, να είμαστε προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για βιομηχανικά έργα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το ποιο θα είναι το όριο στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και αυτό για να μην αποφευθεί σταδιακή πρόοδος, γιατί όταν μιλάμε για βιομηχανικά έργα και βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη ευθύ εξ αρχή, ίσως τότε κινδυνεύουμε να αποκλείσουμε κάποια έργα, κάποια προγράμματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιλεχθεί μεσοπρόθεσμα δεν εμφανίζονται οι θαυματουργές λύσεις εν μία νυχτή. Γι' αυτό και θα θέλαμε να στηρίξουμε σταδιακά προγράμματα με το Invest EU προκειμένου να προωθηθεί παρετέρω η καινοτομία. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες μου. Συμφωνούμε βέβαια με τις κύριες γραμμές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλώς θέλουμε τη στήριξή σας για τη βιωσιμότητα, ε, το κλίμα, την ε, παρακολούθηση και πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την ενσωμάτωση του παράγοντα κλίμα στις διάφορες πολιτικές. Και επίσης όταν υπάρχει καινοτομία με υψηλό κίνδυνο και αυτή πρέπει να στηριχτεί στα πλαίσια του Invest EU. Αυτές είναι οι προτάσεις μου λοιπόν και προσβλέπω στις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των σχεδόν εισηγητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οι σχεδόντες εισηγητές, οι εισηγητές πρώτο ο κύριος Γραμματικάκης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να επενέσω τον κύριο Μπέλετ για τη γνωμοδότησή του και το έκανε ξεκάθαρο και σήμερα ότι με τις ε, τροπολογίες που ο ίδιος θα εισάγει ε, η όλη προσπάθεια γίνεται ακόμα καλύτερα. Το κυριότερο είναι ότι έχει συνδέσει ο εισηγητής την ε, σχέση ανάμεσα στο Invest EU και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρώπη στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Συγκεκριμένα, για να είμαστε συνεπείς με το στόχο του 30% για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο σύνολο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πρέπει να φανούμε αρκετά πιο φιλόδοξοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχεδιασμό του Invest EU. Δεν αρκεί λοιπόν ο στόχος του 50% να περιορίζεται στον τομέα βιώσιμες υποδομές, ενός μόνο από τους τέσσερις τομείς του Invest EU Σωστά λοιπόν, πολύ σωστά ο εισηγητής προτείνει ο στόχος που σχετίζεται με τις δαπάνες για το κλίμα να καλύπτει ολόκληρο το InvestEU, δηλαδή και τους τέσσερις βασικούς πυλώνες, που όπως ξέρετε είναι οι βιώσιμες υποδομές, η έρευνα και καινοτομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επενδύσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι Πιστεύω όμως ότι πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τους τρεις αυτούς πυλώνες και να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τα έργα που θα θέλαμε να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του τομέα έρευνα και καινοτομία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα που να επιτρέπουν τη διείσδυση της επόμενης γενιάς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπαταριών. Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ανεξάρτητων συστημάτων με ποσοστό διείσδυσης που να φτάνει το 100%. Τέτοια προγράμματα θα ήταν ιδανικά για απομονωμένες περιοχές και ειδικά για τα νησιά που πρέπει νομίζω να μας απασχολούν ιδιαίτερα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η σημασία του InvestEU είναι τεράστια, κυρίως όσο η Τραπεζική Ένωση είναι ακόμα, το ξέρουμε καλά, πολύ ατελής στα κράτη που το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ακόμα σε κρίση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφικτιούν και οι νέοι επιστήμονες, το υπογραμμίζω αυτό, αδυνατούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική στρέβλωση της αγοράς και αυτές ακριβώς τις στρεβλώσεις ελπίζω θα διορθώσει το InvestEU. Τέλος, όσον αφορά τον τελευταίο και μικρότερο πυλώνα, τις κοινωνικές επενδύσεις. Κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να έχουν οι περιοχές εκείνες που εξαρτώνται από οικονομίες υψηλής έντασης άνθρακα. Πρέπει να δώσουμε στις περιοχές αυτές την ευκαιρία να προσαρμοστούν στη νέα αυτή εποχή. Κύρια μέρημνά μας, και νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι, πρέπει να είναι ότι η μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η πολύ σπουδαία αυτή μάχη, δεν πρέπει να οδηγήσει κανένα εργαζόμενο σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. κύριο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με την σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή οι αρχικές μου παρατηρήσεις ακολουθούν τη γραμμή της Επιτροπής και πιστεύω ότι ο κύριος Μπέλετ εισήγε μερικές, ε, μερικά στοιχεία που καθιστούν την πρόταση πιο δυνατή. Βλέπω ότι αυξάνονται οι φιλοδοξίες μας σε ό,τι αφορά την επένδυση στο κλίμα. Θα ήθελα να δούμε αν θα μπορούσαμε να το αυξήσουμε περαιτέρω έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε και τα τέσσερα διαφορετικά μέρη του προγράμματος και να κινηθούν προς μία κατεύθυνση, όχι μόνο ένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι χρήματα που επενδύονται για το κλίμα και αυτό δεν ε, θα γίνει ε, ένα μέσο για την πραγματοποίηση πολιτικών φιλοδοξιών. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να συμβάλλουμε σε ό,τι αφορά την βελτίωση την ε, επίλυση των κλιματικών προβλημάτων. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και θα πρέπει να έχουμε την ε, βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα προχωρήσουμε βάσει ορισμένες βασικές γραμμές. Όπως είπε ο κύριος Μπέλετ, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια με βάση διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις πολιτικές μας και να συμβάλλουμε έτσι ώστε οι πολιτικές μας να κινηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούμε να ελέγχουμε πού πηγαίνουν οι επενδύσεις και τι, κλιματικές, ε, ε, τι αλλαγές στο κλίμα επιφέρουν. Έχω έναν προβληματισμό και θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημά μου στην Επιτροπή. Η, το ταμείο αυτό ήταν υπό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι. Τώρα η Επιτροπή έχει αναλάβει αυτή την εξουσία ενδεχομένω. η Επιτροπή έχει πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Θα ήθελα να θέσω όμως ευθέω το ερώτημα γιατί έγινε αυτή η αλλαγή σε ό,τι αφορά την εξουσία. Ε, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι υπό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να έχω την βεβαιότητα ότι οι τροπολογίες που θα υποβληθούν θα είναι της αρμοδιότητας της ΕΝΔΗ ε, από τη στιγμή που επλέκονται αρκετές ε, επιτροπές. Εμείς σας προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε αυτές τις επιτροπές. Ε, η συζήτηση που θα ακολουθήσει στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις δίχως άλλο θα είναι ιδιαίτερα εκτενής. Ευχαριστώ. Κύριε Βυσσινεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η το πρόγραμμα InvestEU θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος προώθησης των επενδύσεων. Οι πόροι που έχουμε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλοι, αλλά δίχως άλλο αυτό οδηγεί σε περαιτέρω ιδιωτικές επενδύσεις. Και θα μπορούσαμε ήδη να θεωρήσουμε ότι έχει στεφτεί από επιτυχία το πρόγραμμα. Ήδη έχουμε εστιάσει την προσοχή μας αυτό που αφορά εμάς. Βεβαίως το βασικό είναι τα θέματα που αφορούν το κλίμα. Η Επιτροπή προτείνει το 50% των πόρων που να δαπανώνται για υποδομές και προτείνει ότι αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Αυτό το κατόφλι είναι πάρα πολύ ψηλό και πραγματικά με προβληματίζει αυτό το θέμα, γιατί πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε τους στόχους μας. Εάν τους συρρυκνώσουμε, αυτό θα σημάνει καταρχάς ότι ορισμένα κονδύλια δεν θα χρησιμοποιηθούν και δεύτερον ότι ενδεχομένως δεν θα κατανεπιθούν με ίσο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης γνωρίζουμε ότι μερικές χώρες μέλη είναι πιο προηγμένες σε σχέση με άλλες σε ό,τι αφορά ενεργειακά θέματα. Και για το λόγο αυτό θα ήθελα να προτείνω να προσεγγίσουμε το όλο θέμα με ένα ευρύτερο τρόπο. Βεβαίως θα πρέπει να περιορίσουμε τις ε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στι κλιματικές αλλαγές. Αλλά εδώ θα πρέπει μεταξύ των άλλων συμπεριλάβουμε ορισμένες πτυχές του κοινωνικού κόστους που αφορά αλλαγέ στην οικονομία. Δεν γνωρίζω αν ξέρετε την έκθεση του, ε, την κοινή έρευνα ε, σχετικά με τις προκλήσεις τις περιοχές εξόριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολύ φιλόδοξε πολιτικέ για το κλίμα ενδεχομένω θα σημαίνουν ότι περιοχέ που έχουν βασίσει την οικονομία του στον άνθρακα θα δουν την ανταγωνιστικότητά του και τι θέσει εργασία να περιορίζονται. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτέ τι περιοχέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα InvestU θα πρέπει να γίνει η βασική πλατφόρμα της υποστήριξης αυτών των περιοχών. Πολλά ε, έχουν υποθεί για αυτές τις περιοχές, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει. Ο κύριος Μπένετ πολύ σωστά ε, είπε ότι ότι η όλη η, διαχειριστική δομή του ε, ταμείου αυτού θα πρέπει να μείνουμε στον προπολογισμό τη ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει κάτι που έμεσα συνδέεται το, με το θέμα και θα πρέπει να συζητηθεί εδώ. Η, το σχέδιο της Επιτροπής ε, δεν κάνει αναφορά στο βασικό ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύω ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να είναι βασική υπεύθυνη για τον καταμερισμό των πόρων για τρεις λόγους. Πρωτίστως είναι έμπειρη. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις ε, ορσιακές πολιτικές. Και τρίτον, και αυτό είναι το πιο βασικό, κινείται, δραστηριοποιείται σε όλες τις χώρες μέλη. Με προβληματίζει λίγο, με ανησυχεί λίγο το ότι τα χρήματα τα που έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορούσαν ενδεχομένως να μην κατανεμηθούν με δικαιοσύνη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των ε, περιφερειών και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να είναι βασικά υπεύθυνη για την κατανομή των πόρων. Η ΕΤΕ έχει μια δική της ε, ε, πολιτική για το κλίμα και νομίζω ότι κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα πρόβλημα με το να συζητήσουμε να αναλάβει αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σεκάουτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι λακωνικότατο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ο Νίλ μου ζήτησε να μην είμαι σύντομο. Οπότε θα τα πω όλα. Δύο σελίδε. Θα είμαι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ τον Ιβο Μπέλε, τον εισηγητή. Ενίσχυσε την ε, πρόταση με αυτά που έκανε ο εισηγητής. Υπάρχουν ένα-δύο θεματάκια πρέπει να καλυφθούν. Ο κύριος Μπελέτ το φροντίζει. Πρώτα απ' όλα, αν δείτε τα τέσσερα παράθυρα που έχουμε εντοπίσει στην πρόταση για το InvestEU, η πρόταση προτείνει να καλύψει μόνο ένα από τα τέσσερα παράθυρα με μέτρα κατά του κλίματος, που αυτό είναι οπισθοχώρη σε σχέση με το ΕΦΣΥ. και έχουμε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο, πολλές επενδύσεις ε, κατευθύνονται προ τα εκεί. Και τώρα είναι ένα βήμα υπαναχώρησης και με εκπλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει. Αυτό δεν ταιριάζει με αυτά που ε, διέδιδαν ε, στις διαπραγματεύσεις ΕΦΣΥ και αυτά που προωθούσαν τότε. Αλλά χαίρομαι που προτείνει ο εισηγητή να καλύπτονται και τα τέσσερα παράθυρα. Και αυτή είναι μια γραμμή που πλήρως υποστηρίζουμε. Μετά υπάρχει και η πτυχή του κλίματος που λάβετε υπόψη. Άρα οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να πηγαίνουν κατά των στόχων καταπολεμήσεως τη αλλαγή του κλίματος που έχουμε θέσει. Επίσης υπάρχει και ένας στόχος που είναι οι επενδύσεις που βοηθούν για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά το κλίμα. Και εκεί ο εισηγητή ισχυροποιεί την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίες εμεί που ανεβάζουν κάπως τον πύχη πιο ψηλά από όταν έχει θέσει ο εισηγητή, αλλά ήδη καλωσορίζουμε το ότι εισηγητή τουλάχιστον βάζει ψηλά τον πύχη, πιο ψηλά από αυτόν που τον βάζει, από τη θέση που τον έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σα εξέπλησε το αντίθετο άλλωστε. Αυτό θα κάνουμε. Και κάτι άλλο. Ο εισηγητή προσπαθεί να τα αφήσει στι αρμοδιότητε Επιτροπή Ένβη, αλλά πρέπει να δοθεί γενικά η προσοχή στην μετακίνηση των επενδύσεων. Κινούνται από κοινοφελεί υπηρεσίε προς συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Είναι μια τάση που είδαμε στα πλαίσια του ΕΦΣΥ, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ένα-δύο προβλήματα πρέπει να καλυφθούν. Πρώτα απ' όλα, τι βλέπουμε, ότι με αυτές τις επενδύσεις το δημόσιο, οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν ένα κίνδυνο. Και αν πάνε στραβά τα πράγματα, πληρώνει η κυβέρνηση. Και όταν υπάρχει κέρδος, ωφελούνται ε, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι και πάντα το συζητούσαμε και στα πλαίσια του ΕΦΣΥ και θα το εξετάσουμε ξανά. Τέταρτο σημείο. Βέβαια, ε, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποια είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα της υποδομές για, τις, για, για, τις, για τους δρόμους, για τα ποδήλατα. Ιδιωτικός φορέας θα διθέσει τα χρήματα. Όχι, γιατί δεν είναι κάτι κερδοφόρο οι αλλά είναι προς το δημόσιο συμφέρον να γίνει. Αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε εκτός και ελοχεύει και άλλος κίνδυνος ότι κάπου θα χαθεί αυτή η πτυχή στην μετακίνηση της κατεύθυνσης των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θα υποβάλουμε κατάλληλες τροπολογίες. Εν γέννη υποστηρίζουμε την κατεύθυνση του ε, εισηγητού, αλλά απλώς θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση. Αυτή ήταν η σύντομη εκδοχή, έτσι. Η σύντομη εκδοχή ήταν αυτή. Το εκτιμούμε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κυρία Εκχάουτ. Η κυρία Σάιπερικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια επίσκεψη στη Κομισιόν, με την Κομισιόν σε μια επαρχία και με τους συναδέρφους εδώ και το πρόβλημα είναι ότι τελικά ξεχνάνε οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Υπάρχουν ε, χρηματοδοτικά μέσα, υπάρχει το ΕΦΣΥ. Πώς φτάνει όμως κανείς εκεί. Υπάρχουν ε, και άλλοι μηχανισμοί, υπάρχει κυκλική οικονομία, στόχοι για το περιβάλλον, ναι. Αλλά πώς τα καταφέρνεις. Αυτό ρωτούν οι επιχειρηματίες. Οπότε πολύ χαίρομαι που τώρα έχουμε κάτι νέο εδώ όταν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χαίρομαι που συμμετέχει. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν γρήγορα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε ακόμα χρόνια. Όχι, όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και υπάρχει και κάτι που λείπει για μένα από εδώ και αυτό είναι η δημόσια υγεία. Ε, στην Ολλανδία έχουμε μία συμφωνία όσον αφορά τον αμίαντο για την κατάργησή του. 50.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτία καρκίνου που οφείλεται στον αμίαντο. Δεν μπορεί να περιμένουμε περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και θα υποβάλω και μια τροπολογία για το θέμα του αμιάντου. Να προσέξουμε το θέμα της υγείας. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω όσο γίνεται πιο γρήγορα να ελοπιθούν όλα αυτά που προτείνονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Λάινεν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να επενέσω τον κύριο Ιβο Μπέλετ για την έκθεσή του. Ανέφερε τα σημαντικά στοιχεία. Το θέμα της βιωσιμότητας όμως. Η αξιολόγηση βιωσιμότητας. Αν αυτή αποβεί αρνητική, θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμα κάποια έργα ή είναι απλώς κάποιος προσανατολισμός που δεν χρειάζεται να το σεβαστούμε. Και συμφωνώ ότι πρέπει να υποστηρίζουμε στρατηγικά προγράμματα. Έχουμε διάφορους κανόνες για τη χρήση τεχνολογίας, να αποφύγουμε εκπομπή διοξιδίου του άνθρακου στην περίπτωση ε, χημικών, χάλιβα, τσιμέντου. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι πτυχές. Και με το παλιό πρόγραμμα είχαν γίνει κάποιες επικρίσεις, δηλαδή ότι δεν ήταν νέα προϊόντα, νέα προγράμματα, αλλά τα χρήματα πήγαιναν σε προγράμματα που ήδη είχαν δρομολογηθεί, όχι για καινούρια. Θα μπορέσουμε να κάνουμε επιλογή, να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς καινούριο πρόγραμμα είναι κάτι που έχει ήδη δρομολογηθεί και παίρνει χρήματα. Ευχαριστώ. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Όχι. Η κυρία Γκέγκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής σας όσον αφορά τον Invest EU. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω όσον αφορά την αύξηση του στόχου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά όσον αφορά την αύξηση που προτείνει ο εισηγητής για τον στόχο για τις υποδομές και γενικά το Invest, 35% πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είναι ένας δύσκολος στόχος, γιατί οι στόχοι για τα τρία άλλα παράθυρα, δηλαδή την έρευνα της μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικές επενδύσεις, εκεί θα είναι δύσκολο να στηριχθούν ε, περιβαλλοντικές επενδύσεις. Για τη μεθοδολογία τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση, θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση αυτή, την αξιόπιστη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων. Θα υπάρξει μια τέτοια ομάδα τις επόμενες εβδομάδες και άρα θα υπάρξει ε, σχετική μεθοδολογία και για την ΕΤΕ. Τώρα για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές, εμείς σημειώνουμε το έτοιμά σας, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κατεξοδότηση πράξης. Έτσι καλώ θα συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσει δίχως άλλο το θέμα. Για τα ζητήματα τώρα που τέθηκαν για τη διακυβέρνηση. Αλλαγές σε σχέση με το πρόγραμμα ΕΦΣΥ. Το ΕΦΣΥ δεν ήταν υπό την ΕΤΕ. Ήταν ε, η ΕΤΕ αποκλειστικά και μόνο εφαρμοστικός εταίρος για να ενισχύεται εγγύηση και να ανοίγεται και σε άλλους εταίρους Τράπεζα Συμβουλίου της Ευρώπης για πραγματογνωμοσύνη, για κοινωνικές επενδύσεις, αλλά και για τις εθνικές ε, βοηθητικές ε, τράπεζες. Ο λόγος ήταν να ενισχυθούν όλες οι περιφέρειες και οι επενδύσεις να είναι πιο ε, υπέρ της περιφέρειας και του τοπικού παράγοντα από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Άρα στηρίζοντας μικρά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν και εθνικές τράπεζες να αναλάβουν. Αυτό που μας ενδιέφερε λοιπόν ήταν ε, το άνοιγμα στην εγγύηση. Αλλά αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ως ρυθμιστής πρέπει να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εξηγεί τις αλλαγές που προτείνουμε τώρα στη διακυβέρνηση σε σχέση με το ΕΦΣΥ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Μπέλετ τώρα. Εσείς λοιπόν για να συνοψίσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους. Πράγματι, η βιωσιμότητα. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει συμφωνία από όλου για τη βιώσιμη υποδομή. Έτσι κι αλλιώς θα θέλουμε και τα τέσσερα παράθυρα. Όπως είπε και ο κύριος Πέτρελ εξάλλου στην αρχή, ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου μέσου είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και να είναι πιο εύκολο να υποβάλει κανείς αίτηση για να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Εξού και καινοτομίε ε, στις αλλαγές. Συμφωνούμε. Εκφράστηκαν ανησυχίες Πραγματικά για τη διακυβέρνηση, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έδωσε κάποια επιχειρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δηλαδή επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη. Πρέπει να το συζητήσουμε με τους σκιώδει ηγητέ για να δούμε κατά πόσο πείθουν τα επιχειρήματα τη Επιτροπής, κατά πόσο μας καθησυχάζουν αρκετά ή μήπω θα έπρεπε να υποβάλουμε ε, κάποια τροπολογία όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Invest EU. Άκουσα επίσης και τις ανησυχίες του συναδέρφου του κύριου Γραμματικάκη αλλά και της κυρίας Βυσνιέσκα όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Ναι, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και μας... δεν είναι βέβαια το μεγαλύτερο παράθυρο ε, από τα τέσσερα, αλλά συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους και σίγουρα θα πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο και πρέπει να βρούμε κοινό τόπο για να τονίσουμε τη σημασία που έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ο κύριος Λάινεν αναφέρθηκε στο στοιχείο της παρακολούθησης κατά πόσο είναι ένα κριτήριο soft ή όχι. Όχι, δεν πρέπει να είναι soft, πρέπει να είναι hard πράγματι και δεν πρέπει να αγνοείται κάθε φορά που μπορούμε να υλοποιήσουμε το κριτήριο αυτό, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να είναι ένα soft, κάτι δηλαδή που να είναι στην ευχέρεια του καθενός και να μπορεί και να παραβλεφθεί. Όχι. Άκουσα και την κυρία Σνάιρερ και την πρότασή της για το θέμα της υγείας και τον αμίαντο. Όντως θα μπορούσε κάλλιστα στο δεύτερο παράθυρο να συμπεριληφθεί ε, και κάτι για αυτό το θέμα. Οπότε θα συμφωνήσω με την τροπολογία της πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην ε, συνεργασία μας στο μέλλον. Πρόεδρος, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 9 ε, Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Θα ψηφίσουμε στις 12 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. So the first vote λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία Λοιπόν, ωραία πρόταση οδηγία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2004-37 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που έχουν σχέση με ε, έκθεση σε καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα στο χώρο εργασία. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική πρόταση 4 και 7. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε κάθε τροπολογία. Τροπολογία 24 και 10. 25 και 10 μαζί ψήφι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται 28, 11 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 12 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεκα... παρακαλώ για να σας ακούσω. Η συμβαστική πρόταση 2. Θέλετε να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Το, το, το, το ξέρετε όμως ότι ψήφισε κατά. Α, ωραία. Να ελέγξουμε τη συμβαστική προς 2. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική πρόταση 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά Α, την έχουν αποσύρει. Συμβαστική πρόταση 5 υπέρ. Εντάξει. Τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Είναι και ζαβό αυτό. And it is rejected. Madame Mellin, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι μόλις παραστήκαμε σε μία καρικατούρα της δημοκρατίας. Θέλησα να ευχαρι... Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές που σε αυτό το κείμενο που ήταν τη Επιτροπή και που απλά και μόνο έφερε το όνομα του εισηγητή. Θα ήθελα να πω ότι μιλάμε για τα συμφέροντα, ε, αλλά εδώ μιλάμε για το εργαζομένο, αλλά εδώ μιλάμε για μία παροδία Τρίτη φορά μιλάμε για αυτή την έκθεση που έχει υποβληθεί από την ομάδα μας. Αυτό θα αποστερήσει την Επιτροπή Απασχόρησης από τη γνωμοδότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και αν αναφέρουμε τον αριθμό των πραγματικών και δυνητικών θανάτων που οφείλονται σε επαγγελματικού λόγους θα μιλάμε για 6 εκατομμύρια σε 60 χρόνια. Κάτι που περιφρονούμε και παρατηρώ ότι μερικοί από τους συναδέλφους φαίνεται, φαίνεται ότι δεν ακούνε καλά, δεν το έχουν προσέξει καλά και θεωρούν ότι μερικοί θάνατοι ελέγχονται καλύτερα από τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ψηφοφορία... χρήση για, ε, της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς, ε, συμβαστική πρόταση 1, υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 42 ε, υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται, 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική πρόταση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πρόταση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 ε, ε, υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά αρχής ψηφοφορίας. Να δω το ΕΛΚ. Φρανσουάζ. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογή 68 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7 υπέρ κατά αποχές υπέρ μισό λεπτό να ελέγξουμε. Συμβαστική πρόταση 7 αρχής ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ελέγχουμε την 76 Πέραση στις πληροφορίες απορρίπτεται Συμβαστική πρόταση 8. Υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να για να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Αρχή ε, της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Για να ελέγξουμε, για να ελέγξουμε. Το 84. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ε, ε, με συγχωρείτε, συμβαστική πρόταση είναι υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική πρόταση 10 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε παρακαλώ. Ε, Ψήφι υπέρ, κατά, από το το, το 13-14 ε, υπέρ κατά για να ελέγξουμε το 14 ελέγχουμε το 14 πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται συμβατική πρόταση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4, η πρόσβαση 14 υπέρ κατά εγκρίνεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική πρόταση 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας.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 ε, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος για την 29 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 29 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 34 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 34 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 51, όχι, ναι, 51 υπέρ, συγγνώμη, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 54 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Για τη 2 ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Wow. Μία αποχή και μόνο. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Κάποιοι από εσά μπορείτε να αποχωρήσετε ησύχω από τη συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο στην Ολομέλεια. Έχουμε ακόμα ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση επιτροπολογιών για διαφάνεια και βιωσιμότητα τη αξιολογήσεω κινδύνου πλευρά Ευρωπαϊκή νόσων στην αριστεία τροφίμων. Η κυρία Ζόμερ είναι η συγχύτρια. Θα τη δώσω παρευθύ το λόγο αφού επικρατήσει κάποια ησυχία στην αίθουσα. Help us keep the voice down. We are nearly there. Shh. Κύριε Σόμερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, πράγματι, πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την αναθεώρηση κανονισμού Εμένα μου έκανε εντύπωση που είχαμε ήδη 539 τροπολογίες μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Βέβαια προς το παρόν έχουμε τις τροπολογίες μόνο στα αγγλικά από σήμερα το μεσημέρι και δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι πρόλαβαν να μελετήσουν όλες αυτές τις τροπολογίες, φαντάζομαι πως όχι, ηρωνικά το λέω. Στους σκιώδες συζητητές θα το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέρφους, οι οποίοι αποφάσισαν να αντιδράσουν σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, από το κόμμα μου ήδη έχουμε κάποιες τροπολογίες για το μέλι και για την προέλευσή του. Οπότε θέλω να ζητήσω από την Πρόεδρο να τις αποσύρει αυτές τις τροπολογίες γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κανονισμό το θέμα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, κυρίως όταν πρόκειται για την εκτίμηση κινδύνου και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Οι χώρες μέλη δεσμεύτηκαν ε, πάντως να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης που γίνεται. Έρχομαι τώρα στο θέμα του ορισμού εμπειρογνωμόνων στα διάφορα πάνελ, τα επιστημονικά πάνελ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι χώρες μέλη πρέπει να υποβάλουν μία υποψηφιότητα, ένα όνομα. Ε, νομίζω ότι δεν συμφωνεί κανείς μας με αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί θα κόστιζε πάρα πολύ αν ένας από κάθε μία από τις 28 χώρες έπρεπε, αν η κάθε χώρα δηλαδή θα έπρεπε να βρει έναν υποψήφιο, θα κόστιζε πολλά και θα ήταν μεγάλη γραφειοκρατία. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει έπειτα να καλύπτουν όλους τους τομείς. Πιστεύω ότι θα κόστιζε πολύ μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση για τον ορισμό των ε, εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά τώρα τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΣΑ. Πιστεύω και εδώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Εγώ προσωπικά έχω υποβάλει τροπολογίες, έχω δεχτεί τις τροπολογίες κάποιων συναδέρφων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να στείλει δύο εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ. Τουλάχιστον δύο. Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω έκθεση για αυτό το θέμα. Όταν μας ζητήθηκε είχαμε ελάχιστη προθεσμία και δεν προλάβαινα. Επίσης, πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή θέση στο Διοικητικό αυτό Συμβούλιο. Τελικά πόσους θα στέλνουμε. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Οι σκιώδες συγητές θα το συζητήσουμε μεταξύ μας. Τώρα οι μελέτες αντικτύπου για αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες μέλη μπορούν να έχουν το δικαίωμα και οι μεν και οι δε να αναθέσουν τέτοιες μελέτες, να ζητήσουν τέτοιες μελέτες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Πιστεύω όμως ότι τέτοιες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες μέλη δηλαδή και στο Συμβούλιο Υπουργών πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Γιατί αν δεχτούμε την απλή πλειοψηφία για τέτοια θέματα, Θα ακούσουμε πάρα πολλέ επιθυμίες να εκφράζονται για την εκπόνηση μελετών. Έχει νόημα. Ε, τελικά είναι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος που πληρώνει. Τι νόημα έχει να παραγγέλουμε και άλλες μελέτες αξιολόγησης, ενώ έχουμε τόσες μελέτες που συσσωρεύονται πάνω στα γραφεία μας. πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό. Οπότε λέω ότι για να ζητήσει κανείς ε, μελέτη θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη. Να μπορούν να το συζητάνε μεταξύ τους για να αποφασίσουν. Ένα άλλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αν όλα τα όργανα μπορούν να ζητήσουν την εκπόνηση τέτοιων μελετών και με απλή πλειοψηφία μόνο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι θα καταλήγαμε σε πολιτικοποίηση των διαδικασιών. Δεν θα έπρεπε. Είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Και τελειώς κινδυνεύουμε να διονύζουμε τις διαδικασίες για την ε, άδεια. Ε, συνάδελφοι έχουν προτείνει τροπολογίες που μιλούν για την εφαρμογή της σύμβασης του άρχους. Όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά ζητήματα. Διάφοροι συνάδελφοι μου μίλησαν ε, γι' αυτό όταν πριν το καλοκαίρι είχα παρουσιάσει ε, το σχέδιο εκθεσής μου. Υπάρχει συνεπώς ένα έγγραφο τοποθέτησης από μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με το περιβάλλον. Που λέει ότι δεν πρέπει να βασιστούμε στην σύμβαση αυτή του άρχους για να ψηφίσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Είναι αναγκαίο αυτό. Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, επίσης, οι οποίες θέλουν να απαλληφθεί η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μα είναι παράδεκτο κάτι τέτοιο. Γιατί τα πνευματικά δικαιώματα είναι δικαιώματα. Δεν βλέπω γιατί στα πλαίσια αυτού του κανονισμού να μην ε, εφαρμόζονται. Οπότε, ότι δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των προϊόντων, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα γι' αυτό, μπορεί να βγει, κατά τη γνώμη μας. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες από τις συμβουλευτικέ συζητήσεις που γίνονται. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ευρύ. οι προπαρασκευαστικέ συναντήσεις γίνονται για να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξέρουν πώς μπορούν να υποβάλουν αιτήσει στην ΕΦΣΑ για να μην μπερδεύονται με το τι έγγραφα πρέπει να υποβάλουν ή τι λεπτομέρειες μπορεί να λείπουν από τις αιτήσει τους. Οπότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις άπαξ και φοβούνται ότι η τι λεπτομερειες μπορει να λειπουν απο τις αιτησει τους οποτε οι μικρομεσαιες επιχειρησει απαξ και φοβουνται οτι η δημοσιευση ε, των στοιχείων θα έχει σαν αποτέλεσμα να μάθει ο κόσμος όλος τα μυστικά τους, δεν θα συμμετέχουν καν. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι που δημιουργούν απασχόληση. Αν όμως αυτές οι μικρομεσαίες βρίσκονται αντιμέτωπες με εμπόδια, τότε έχουν ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα το ιδιαίτερο επίμαχο θέμα είναι το πότε πρέπει να δημοσιεύονται τα πιο ευαίσθητα στοιχεία. Και υπάρχουν εδώ πέρα δύο ομάδες, δύο στρατόπεδα. Κατά τη γνώμη μου, πριν από το καλοκαίρι, συζητούσαμε το περιεχόμενο των συμβουλευτικών συναντήσεων και των αιτήσεων που θα έπρεπε να δημοσιεύονται όλα όταν υποβάλλεται το αίτημα. Ε, ο φόβος είναι ότι οι ιδέες τους μπορεί να φτάσουν σε χέρια ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να τους κλέψουν τις ιδέες. Αν οι πληροφορίες αυτές της καινοτομίας υπάρχουν στο αίτημα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς για ποιο προϊόν πρόκειται. Και όσο πιο πολύ κρατάει η αδειοδότηση, που σε εμά πολλές φορές κρατάει πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες, μερικές φορές δεν περνάει καθόλου χρονικό διάστημα αλλού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται για την αδειοδότηση πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μπορεί από άλλες αγορές να ξεπεταχτούν τέτοια προϊόντα κλέβοντας τις ιδέες των δικών μας. Οπότε δεν θα είναι επιτυχία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν επενδύσει και τελικά κάποιος άλλος θα υποφεληθεί για αυτό το προϊόν. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης στη διαφάνεια και στο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες. Ας δούμε και την ε, υπηρεσία φαρμάκων. Εκείνοι πότε δημοσιεύουν τις πληροφορίες. Πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με αυτούς. Οπότε αν δείτε τις νέες τροπολογίες θα δείτε ότι προσπαθώ να λάβω υπόψη μου τις ιδέες άλλων συναδέρφων. Έτσι λοιπόν τώρα προτείνω πληροφορίες τη στιγμή της δημοσίευσης του σχεδίου γνωμοδότησης γιατί πρώτα έρχεται ένα σχέδιο γνωμοδότησης, μετά γίνεται η διαβούλευση. Και μετά οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν αν λείπει κάποια μελέτη ή κάτι και όταν τελειώσει η διαβούλευση, τότε η ΕΦΣΑ μπορεί να υποβάλει μια τελική γνωμοδότηση και να την δημοσιεύσει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ήδη η ΕΦΣΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων. Οπότε, χωρίς να έχει την υποχρέωση. Έτσι, πάντως, αυτή η περίοδος διαβούλευσης οδηγεί στο να αλλάξουν την τελική τους γνωμοδότηση σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης. Είμαι υπέρ της διαφάνειας, μεν, αλλά δεν θέλω να πληγούν έτσι διάφορες επιχειρήσεις όπου θα δουν να δημοσιεύονται οι πληροφορίες τους πρόωρα. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. Η ΕΦΣΑ να ετοιμάζει μια προκαταρτική δημοσίευση, θα το εξετάζουν αυτό οι ενδιαφερόμενοι στην περίοδο διαβούλευσης και μετά, αφού έχει ληφθεί υπόψη η διαβούλευση, η ΕΦΣΑ θα καταλήγει στην άποψή της. Ίσως πάνω σε αυτό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σόμερ που ήταν όντως εκτενής η παρουσίασή σας. Τώρα στρεφόμαστε στους κοιόδες εισηγητές να δούμε ποια είναι απόψη τους. Ο κύριος Πόρτς πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ βεβαίως και την εισηγήτρια για την προσπάθεια που έκανε να επαναδιατυπώσει το σχέδιο. Ακούτε τη μετάφραση? Ωραία. Εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα καλύτερο σύστημα αδειοδότησης που δεν ε, ε, θα είναι ευαίσθητο σε εξωτερικές πιέσεις, ενώ εύκολα θα μπορούμε να εντοπίζουμε περιπτώσεις απάτης. Ε, μερικές παρατηρήσεις. Καταρχάς θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ανεξάρτητους επιστήμονες, χωρίς να χρειάζεται να ζητάμε άδεια, αυτό είναι ο μόνος τρόπος ε, να καταλήξει κανείς σε έγκυρες επιστημονικές γνώσεις και βεβαίως να παράσχει προστασία στο περιβάλλον. Η αναθεώρηση του Γενικού Νόμου για τα τρόφιμα καλύπτει μία σειρά από ξεχωριστά θέματα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της νομοθεσίας που καλύπτεται από τη Συμφωνία του Άρκους, όπως νομοθεσία που αφορά τα, ε, ε, τα μεταλλαγμένα και άλλα θέματα που δεν αφορούν εκπομπές προς το, ε, στο περιβάλλον και εκεί η επέκταση του, της συμφωνίας του Άργου θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικές και αβεβαιότητες. Υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να διασφαλιστούν, αλλά όχι εις βάρος της ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να, βασίζ, να έχουμε μια προσέγγιση που να βασίζεται σε κινδύνους. Πιστεύουμε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ε, δημιουργήσουμε ένα καθεστώς κοινοποίησης και παράλληλα να προστατεύουμε τους από την κλοπή των ιδεών τους από ανταγωνιστές. Σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει καθυστέρηση, δηλαδή σε σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει λόγο, ε, ιδιωτολογία καθυστέρησης θα πρέπει να έχουμε την ε, βεβαιότητα ότι ένα νέο σύστημα κοινοποίηση δεν θα παρεμποδίσει την εισαγωγή νέων προϊόντων. Αυτό αφορά νέες τροφές που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις διαδικασίες στις οποίες αναφέρθηκε η συγκήτρια, τύπος, το όνομα του ετούντος, τύπος της αίτηση και ε, μετά ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι αυτό θα αφήσει χρόνο για μία εξέταση του θέματος και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε ένα σωστό συμβιβασμό σχετικά με αυτά τα θέματα. Okay, thank Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φέντελε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την ε, ε έκθεσή της. Εγώ θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά ο χρόνος πιέζει, ε, θα πρέπει να φύγω και βεβαίως θα πρέπει να βιαστώ. Πιστεύω ότι όταν αύριο το πρωί ξεκινήσουμε τις πραγματικές διαπραγματεύσεις, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το κάνουμε αυτό σε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούνται πιέσεις στην ΕΦΣΑ. Συνεχίζεται μια συζήτηση αρκετές φορές ε, εδώ και ελπίζω ότι θα μπορέσει να μπει κατά μέρο αυτή η συζήτηση και να ασχοληθούμε με τον κανονισμό έτσι ώστε να μην έχουμε ένα θέμα που θα μας απασχολεί διαρκώς. Η ΕΦΣΑ ήταν μια ιστορία επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατάφερε να εξασφαλίσει την ασφάλεια την προστασία των τροφίων για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Όταν ήμουν νέος, αν κανείς πήγαινε στην Ισπανία για διακοπές, το πρώτο πράγμα που του έλεγαν ήταν να μην τρώει αυγά και κοτόπουλο, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος της σαλμονέλας. Ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί κανείς να φάει άφοβα και ένα μελάτο αυγό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι πάρα πολύ, ε, χάρη στη δουλειά που έκανε η ΕΦΣΑ, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα οι συνάδελφοι να έχουν κατά νου ότι η σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων δεν ήταν ποτέ καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι πραγματικά γλίτωσε πολλούς ανθρώπους ε, από πολλά δεινά και πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να ζήσουν πολύ περισσότερο χάρη σε, ε, αυτές τις ε, προβλε... Ε, σε αυτά τα μέτρα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας, που θα πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή. Τι πρέπει να είναι διαφανές, τι θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο κοινό. δεν έχουμε σκοπό να αποκρύψουμε πληροφορίες από τους πολίτες για θέματα κοινοποιηθούν νωρί ενδεχομένως θα κλαπούν από κάποιον άλλον, από κάποιον ανταγωνιστή. Και αυτό θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την εξέλιξη της καινοτομία στον τομέα. Θα πρέπει βεβαίως τη δια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης να τονίσουμε ότι μειώνονται οι καινοτομίε στον τομέα των τροφίμων και αν ε, νομοθετούμε καθ' υπερβολή ε, θα χρειαστεί περισσότερος χώρο και πάρα πολλέ εταιρείε ενδεχομένω θα εγκαταλείψουν την ήπειρό μα ε, προ όφελο άλλων, αλλά θα είναι μία απώλεια για την Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Στην ε, συζήτηση για το πολιετές ε, πλαίσιο διεξάγεται και μια συζήτηση για το πόσα χρήματα θα πρέπει να δοθούν στην ΕΦΣΑ, γιατί η ανεξαρτησία της έρευνας είναι σημαντική και θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την ε, έρευνα και ότι βασίζουν εκεί την κρίση τους. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε τις τροπολογίες αυτές με έναν τρόπο φιλικό. Η, ε, η συγγήτρια έκανε παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να, να με βρουν ε, σύμφωνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα Κάτι που θα τονίσω κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διεξαχθεί μία συζήτηση επιδεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν μιλάμε για τρόφιμα και ασφάλεια τροφίμων. Θα πρέπει να βασιζόμαστε σε πρακτικές διαδικασίες που έχουν αποδειχθεί λειτουργικές και που στηρίζονται από την κοινότητα των ερευνητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που ανησυχώ ότι σας παραπλανήσατε όταν ήταν νέος για την Ισπανία. Φοβούμαι ότι ίσως αυτό να επηρέασε και τις εργασίες σας στο Κοινοβούλιο. Τι σας κάνανε όταν σας ήταν μικρός. Η κυρία Χάζενκαμπ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις της κυρία Σόμερ όσον αφορά αυτή την ευαίσθητη έκθεση. Προφανώς είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ευαίσθητο, εξού και οι πολυάριθμες τροπολογίε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην συνάδελφο για να τα καταφέρει. Εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, διαφάνεια, από τη μία και αξιοπιστία από την άλλη, και από την άλλη η μεριά επίσης και ανεξαρτησία των μελετών. Γιατί από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, οι πολίτες θέλουν να έχουν πρόσβαση, άρα να υπάρχει διαφάνεια και αυτό πρέπει και εμείς να το εξασφαλίσουμε. Δεν διάβασα βέβαια το αγγλικό κείμενο, των τροπολογιών δηλαδή, αλλά ελπίζω αυτό να ληφθεί υπόψη επαρκώς. Η Επιτροπή λέει ότι είναι προτεραιότητά της να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, πώς θα γίνει αυτό. Οι πολίτες δεν πρέπει να δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο Αντίθετα, πρέπει να τους διευκολύνουμε. Έπειτα και για τον κλάδο και για την ΕΦΣΑ, αν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό θα βοηθήσει τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστατεύει περισσότερο τον κλάδο και όχι το περιβάλλον και τους πολίτες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η αρχή που πρέπει να κυριαρχήσει εδώ πέρα είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων και των ζώων να μπορούν να ζουν με ευημερία. Το δικαίωμα στην υγεία επίσης και της διαβίωσης σε ένα υγιεινό περιβάλλον και αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτά που υπάρχουν ως δικαιώματα και είναι και το Κοινοβούλιο υποχρεωμένο να υποστηρίζει αυτά τα δικαιώματα πάντα. Έπειτα, αξιοπιστία και ανεξαρτησία των μελετών. Έχει μεγάλη σημασία οι μελέτες στην αρχή της διαδικασίας να γίνονται γνωστές, έτσι ώστε και οι επιστήμονες και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μπορούν να κρίνουν αυτές τις μελέτες. Οπότε δεν πρέπει η ΕΦΣΑ ε, να κάνει την διαδικασία αξιολόγησης ε, και κλεισμένο των θυρών. Έπειτα ο κλάδος είναι υπεύθυνο για τις μελέτες που γίνονται όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει να γίνονται μελέτες από ανεξάρτητους επιστήμονες και όχι να επηρεάζονται από την βιομηχανία, από τον κλάδο. Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η έκθεση, να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία που είπα για να αποφεύγουμε φαινόμενα σαν και αυτό της Μοντσάντο και της ε, Γλυκοσφασάτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Χάρσλικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αν το ήξερα, θα μπορούσαμε να είχαμε διοργανώσει μια συνεδρίαση σκιωδών. Μεταξύ μας είμαστε τώρα. Δεν θα αναφέρω τα ίδια αναφερθέντα. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάτι που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στην παρουσίαση που είχε κάνει στην πρωτοβουλία περί Και θα πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και χαίρομαι που το ακούω ότι η σύμβαση του Άρχους που είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί και σύμφωνα με αυτήν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αμφισβητηθούν οι προσεγγίσεις που θα ακολουθηθούν. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες, τις υποβάλαμε πριν από τις θερινές διακοπές. Το άρθρο 39 μας προβληματίζει, το άρθρο 39 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί λέει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η προσέγγιση σε λιγότερο άνοιγμα από ότι περισσότερο, λιγότερη διαφάνεια. Πώς το δικαιολογεί αυτό. Στη συζήτηση μιλήσαμε για συμφέροντα εταιριών, για συμφέροντα του δημοσίου και πού μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό. Πρέπει να σταθμίσουμε την κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί κατάσταση κατά την οποία τα συμφέροντα των επιχειρήσεων θεωρούνται πιο σημαντικά διότι εδώ παίζεται η αξιοπιστία του ΕΦΣΑ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η αξιοπιστία. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί καχυποψία. Διαφορετικά είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Και θέλαμε πριν το καλοκαίρι να ξέρουμε πότε θα δημοσιευτεί το κείμενο. Αυτό θα ήταν ένα βήμα πρόοδου Πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέλος μιας διαδικασίας, να έχουμε φτάσει στο τέλος και τότε να συμμετέχει η ΕΦΣΑ. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη καχυποψία εκείνων που δεν συμμετέχουν άμεσα στις συζητήσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σημειωθεί πρόοδος πρέπει να το κάνουμε δεν πρέπει να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση αντίθετη από τη Θα ήταν προβληματικό κάτι τέτοιο. Πρέπει να εμπλακεί και κοινή γνώμη πιο πριν σε αυτά που κάνουμε. Τι γίνεται με τα, με τα μυστικά των επιχειρήσεων, τις επιστευτικές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι κάποιες επιχειρήσεις, κάποια επιχειρηματικά μυστικά προστατεύονται για λόγους ε, ανταγωνιστικότητας ανταγωνιστικότητα εν συγκρίση με επιχειρήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε όμω και τη χρυσή τομή. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Για την ΕΦΣΑ αυτή καθ' αυτή καλωσορίζω το ότι λέτε ότι έχουμε δύο εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου που θα συμμετέχουν, αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Τι γίνεται όμω με τον διορισμό των επιστημόνων. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει η διαδικασία σχετική να είναι διαφανής. Αν δεν έχουμε πιστήμονες στο πάνελ, αλλά εκπροσώπους των αρχών, αυτό δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τις αρχές, πώς βλέπει ο κόσμος τις αρχές, την, το φορέα αυτό μάλλον, πώς εξασφαλίζουμε ε, τι γίνεται με τις μελέτες εξακρίβωσης. Και κάτι άλλο, η χρηματοδότηση αν πρόκειται να γίνει εξακρίβωση μιας μελέτης. Τότε πρέπει να διατεθούν και τα κατάλληλα χρήματα. Γιατί να πληρώνει ο φορολογούμενος. Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα φορέα που θα έχει μια χρηματοδότηση και από αυτά τα χρήματα θα πληρώνονται οι μελέτες. Έτσι θα εξασφαλίζουμε ότι η ΕΦΣΑ έχει αρκετά ε, χρήματα να κάνει τις αναγκαίες εξακριβώσεις σχετικά με τις μελέτες. Θα ήταν μια καλή λύση αυτή. Και θέλουμε να είμαστε όσο πιο θετικοί γίνεται απέναντι στο κοινό. Να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Ελπίζω αύριο στη συνεδρίασή μα να πετύχουμε κάποια πράγματα, να συμβιβαστούμε, να πετύχουμε κάποια πρόοδο. Ε, Προφανώ θέλουμε να ολοκληρωθεί το ζήτημα αυτό πριν τι επόμενε ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλου πέντε ομιλητέ έχω. Παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε όμως. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν θα θέσω και χρονόμετρο και όριο. Σας Η κυρία Αγίουσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Πρώτον, συγχαρητήρια στην κυρία Σόμερ. Συμφωνώ με όλες τις, τις προτάσεις. Οπότε το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από την εμπειρία ξέρουμε ότι ο κανονισμός αυτός χρειαζόταν μια πιο μεγάλη αλλαγή και πιο πλήρη και όχι να ασχοληθούμε μόνο με την διαφάνεια κλπ. Γι' αυτό και έχω υποβάλει τέσσερις τροπολογίες που παρόλο που δεν αποτελούν μέρος των αλλαγών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικές αλλαγές που προτείνονται. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κοινή διαδικασία όταν υπάρχει κίνδυνος για να κρούμε τον κόνδωνα του κινδύνου. Όταν υπάρχει κρίση, όπως έχουμε με με κάτι άλλο, πρέπει να υπάρχει διαδικασία ε, και εναρμονισμένη μάλιστα και προδιαγραφές κοινέ για όλες τις χώρες μέλη. Επίσης, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην διαχείριση και στην επικοινωνία σε περίπτωση τέτοιων κρίσεων. Όχι όπως τώρα με το σύστημα που έχουμε σήμερα που αποτελεί απλώς ένα εγχειρίδιο στήριξης. Επίσης, πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο ε, τις υποχρεώσεις που έχει η ΕΦΣΑ, που πολλές από αυτές δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των τροφίμων τα θέματα των ιστανίων των φυτών, για παράδειγμα, δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων. Αν μια τομάτα έχει κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί ασθένεια, αλλά δεν επηρεάζει καθόλου την ασφάλεια τροφίμων. Στο θέμα όμως της υγείας των ε, ζώων. Λοιπόν, από τα φυτά καμία ασθένεια, έτσι, οπότε η δεν θα έπρεπε να ασχολείται, να μην ξοδεύει ούτε χρήματα, ούτε προσωπικό για προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα φυτογενομικά των φυτών, γιατί δεν επηρεάζουν καθόλου τη διατροφική ασφάλεια. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με ε, τα ζώα. Δεν ε, πρόκειται μόνο για απλά ζητήματα. Ο, η πανόλη των χείρων, για παράδειγμα, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. εγώ έχω μία επιστολή από τους Ισπανούς παραγωγούς, οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί η ΕΦΣΑ έχει οργανώσει μια ε, διάσκεψη για το θέμα της πανόλης ε, των χείρων της Αφρικανικής Πανόλης. Όταν όμως βλέπει ότι ασχολείται με αυτό η ΕΦΣΑ, σημαίνει ότι όταν εκδηλωθεί σε μία χώρα, τότε η κατανάλωση χείρου κρέατος θα μειωθεί πάρα πολύ, γιατί κάνει τη σύνδεση στο μυαλό του ο καταναλωτής χωρίς να πρέπει. Έπειτα νομίζω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε αυστηροί, αλλά να μην δημιουργούμε ανησυχία στην κοινή γνώμη για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τροφίμων. Η προστασία των ζώων, η ευημερία των ζώων, ούτε και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια των, ε, ε, τη διατροφική ασφάλεια. Οπότε να απαλλάξουμε την ΕΦΣΑ από αρμοδιότητες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφική ασφάλεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Αντελέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την κυρία Ρενάτα Σόμερ, τη συνάδελφο τη δουλειά που έκανε. Οι συμπολίτε μα όλο και περισσότερο διαρωτώνται για το περιεχόμενο του πιάτου του, οπότε υπέχουμε καθήκον να εξασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίε εγκρίσεω φυτογενομικών προϊόντων των τροφίμων να είναι κάτι διαφανέ και ασφαλέ και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και των παραγωγών και των καταναλωτών. επενθυμίσω ότι η Ευρώπη έχει τους, μία από τις ελεγκτικές διαδικασίες τις πιο προθυμένες στον κόσμο όσον αφορά τα φυτοϊγειονομικά προϊόντα και αυτό το κείμενο ακόμη φορά θα κάνει την Ευρώπη πρόδρομο, ε, θα είναι στην πρώτη γραμμή στον αυτό το θέμα. Να υπογραμμίσω ε, ένα λάθος στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Πώς μπορούμε να εισάγουμε από τέτοιες χώρες προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που επιβάλλουν σε αυτούς μα όσον αφορά την υγεία και όσον αφορά το περιβάλλον. Γι' αυτό κατέθεσα τροπολογίες για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών επιβάλλοντας το ότι οι, οι συμφωνίες εμπορικές μεταξύ κρατών και των χωρών θα υποχρεώνουν τι χώρε να πληρούν προδιαγραφέ δικέ μα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία για καλύτερη προστασία της υγείας των συμπολιτών μας. Γι' αυτό θα ήθελα αρχή της κοινοτικής προτίμησης να εφαρμόζεται σε όλους αυτούς τους τομείς, για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την σπουδαία δουλειά που έκανε Κοινάζοντα και τι το διαπιστώνω κοιτάζοντας τροπολογίες και στο πρωτότυπο. Το θέμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε ένα θέμα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που εκ των πραγμάτων υπάρχουν στο εμπόριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είχαν ποτέ αρνητικέ επιπτώσεις και ποτέ δεν τέθηκε υπό συζήτηση η ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό αφορά τα ανθρακοινόνια που ε, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να τεθούν εκτός αγοράς. Γιατί η γνωμοδότηση αυτή δεν βασίζεται στα ίδια τα μόρια, αλλά στην ουσία βασίζεται σε παρεμφερή συνθετικά μόρια και μετά μεταφέρεται στα φυσικά μόρια. Αυτό όμω είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν εκτός εμπορίου ορισμένες ουσίες που βρίσκονται στη φύση και χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Εννοείται ότι έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε να μην συμβούν και πάλι τέτοιου είδους πράγματα. Ένα άλλο θέμα αφορά την ε, διαφάνεια. Αυτό ε, επί αυτού του θέματος ε, έχω ε, υποβάλει μερικές τροπολογίες και επίσης να οι υπόψη από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάιπεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συνάδελφα από το ΕΛΚ που έλαβε υπόψη της, τις παρατηρήσεις μας και θα ήθελα οι επιτροπέ Ελής και να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις της κυρία Σόμερ. Όντω η διαφάνεια πρέπει να είναι αναλλαγική και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι ο κλώδος θα έχει εμπιστοσύνη στην ομοθεσία που προτείνεται και δεν θα επιτραπεί σε ακραίους να μας κατηγορούν για το θέμα της ασφάλειας τροφίμων η ασφάλεια που έχουμε στην Ευρώπη είναι καλύτερη στον κόσμο και δεν πρέπει να εμποδίζεται από τη γραφειοκρατία ή από ανταγωνιστές μας, Κινέζους κλπ. που δεν τηρούν αυτά που πρέπει. Προσοχή λοιπόν πώς θα χειριστούμε το ζήτημα. Υποχρέωση της ιχνολάτησης και της διαφάνειας πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αναλαμβάνουν οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε φορά που γίνεται κάποια αναγγελία, αυτή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να γίνεται κατανοητή σε όλες τις χώρες. Αλλιώς, εφόσον δεν υπάρχει εναρμόνιση, τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά που θέλουμε. Η ΕΦΣΑ είναι πολύ σημαντική. Οι επιστημονικές μελέτες τώρα και οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να δίνονται με τέτοιο τρόπο που να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα. Αλλά βέβαια κίνδυνο είναι ότι οι ανταγωνιστές θα ενημερωθούν για στοιχεία, για καινοτομία, για νέα προϊόντα ή νέες ε, διαδικασίες παραγωγής. Το άρθρο 38.1 και το, ο κανονισμός 78002 πρέπει να λέει ποια θα πρέπει να είναι η δομή. Πρέπει να υπάρξει καλή ισορροπία ανάμεσα στην πληροφορία και να γίνει διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία γενικά και την πληροφορία που δίνεται πριν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της η ΕΦΣΑ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρίσκονται με μειονέκτημα. οι ετούντες θα πρέπει να οργανώνονται κατάλληλα. Thank you. Madam Uh, Κυρία Γκέρλινγκ, ευχαριστώ. Έχω ερώτηση για την εισηγήτρια. Στην αρχική παρουσίαση και στις αρχικές εκθέσεις αναφέρθηκε στην έλλειψη αξιολογήσεως αντικτύπου, διαβάζοντας την έκθεση για να υποβάλω σχετικά τροπολογίες, συνεπέρανα ότι ίσως θα ήταν δυσανάλογο να γίνει αυτό, διότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν επίμαχες. Και είχαμε και καλές προτάσεις της εισηγήτριας. Κάποιοι εξέτασαν λεπτομερώς τροπολογίες, εγώ όχι. Κάποιες τροπολογίες αναφερόταν στη διαφάνεια και αυτό θα συνεπαγόταν ε, αλλαγή της θέσης μας. Η συγγήτρια πιστεύει ότι πρέπει αυτό το τμήμα να εξετάσουμε και να ζητήσουμε αξιολόγηση αντιχτύπου. Δεν πρέπει να κάνουμε σημαντικές, σημαντικές αλλαγές αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάντα τα καταφέρνουν. Αν είμαστε όμως σοβαροί να βρούμε προϊόντα προστασίας των φυτών που βλάπτουν ελάχιστα το περιβάλλον, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό αν δεν προστατεύσουμε την ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα. Και θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει, τότε το λόγο δίνω στον κύριο Σκάνολ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τους κοιόδης εισηγητές και τα μέλη του Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο για την ε, σκληρή δουλειά που έκαναν σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση. Καταλαβαίνουμε τον κατεπήγοντα χαρακτήρα αυτής της ε, πρότασης. Ε, ο χρόνος πίεσε, παρόλο που αυτό δεν μας ικανοποιεί, αλλά θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά και να και δυστυχώς δεν είχαμε την πολυτέλεια να ξοδέψουμε χρόνο για μία αξιολόγηση των επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση αυτή εσιάζεται σε συγκεκριμένα σημεία και δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε μία τέτοια αξιολόγηση συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Νομίζω ότι τη λαμβάνοντας ε, υπόψη τα όσα εισηγητέ, ε, η Αυστριακή Προεδρία έκανε θαυμάσια δουλειά, έκανε διαπραγματεύσει με άλλε χώρε μέλη και πραγματικά έχει επιτευχθεί πρόοδο. Και πραγματικά θα μπορούσα να κάνω παραλληλισμού με, τη, με τα, με τα θέματα που συναντώνται στο Κοινοβούλιο και στην αίθουσα αυτή συγκεκριμένα. Έχουν τεθεί διάφορα θέματα. Συζητήθηκε για παράδειγμα το θέμα της κοινοποίηση των κινδύνων και σε σχέση με αυτό το θέμα συζητήθηκε το θέμα συγκεκριμένων προτάσεων η Επιτροπή δεν είχε επισέλθει δεν σε λεπτομέρειες στην πρόταση. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι είχαμε, υπάρχουν προ, ε, ε, προτάσεις στη διαδικασία επιτροπολογίες και στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινοποίηση των κινδύνων αναγνωρίζουμε ότι είναι βασικό στοιχείο της ενεργικής ανάλυσης κινδύνων και πραγματικά διεισδύει στην όλη διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων και όντως παραδεχόμαστε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, και αυτό είναι σαφές ε, στην ίδια την ε, πρόταση. Όντως υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό για να σταλεί ένα πιο έντονο μήνυμα στις χώρες μέλη για το πώς κοινοποιούνται οι κίνδυνοι γιατί στους πολίτες δεν αρέσει να ακούν αντικρουόμενες γνώμες από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία τους. Ένα άλλο θέμα που αναφέρατε αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει στο να δώσουμε στις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τον ορισμό των επιστημονικών, ε, ε των ε, η ΕΦΣΑ αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες και αυτό υπάρχει και στα διάφορα ιδρύματα των κρατών μελών. Με το πέρασμα του χρόνου όμως δεν θα είναι ε, διατεθειμένοι να ε, απασχολήσουν αυτούς τους εμπειρογνώμονες. Καταρχάς θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τους εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να ζητήσουμε από τις ίδιες τις χώρες μέλη να δώσουν στην ΕΦΣΑ μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης. Βεβαίω, θεωρούμε ότι ο εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΦΣΑ θα συνεχίσει να διατραματίζει κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των κενών σε ό,τι αφορά την πραγματογνωμοσύνη των, από πλευρά των κρατών μελών και θα κάνει μια προσπάθεια να καλύψει αυτά τα κενά. Σε ό,τι αφορά θέματα διαχείρισης θα ήθελα να πω ότι περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ε, ε, ε, εδώ το θέμα είναι η διαχείριση της, της ΕΦΣΑ. Δεν είναι το θέμα της αξιολόγησης των κινδύνων. Μιλάμε για μια λειτουργική συνεδρίαση που συζητάμε θέματα που αφορούν τον προπολογισμό, στρατηγικά θέματα, αλλά όχι το θέμα της αξιολόγησης των κινδύνων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για να σας διαβεβαιώσει ότι οι προτινόμενες αυτές δομές δεν θα παρεύουν στην ανεξαρτησία των επιστημονικών πάνελ. ό,τι αφορά το μοντέλο που επιλέξαμε είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται για όλους τους φορείς. Η ΕΦΣΑ στην υπάρχουσα δομή της αποτελεί την εξαίρεση των κανόνα. Και αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να συμπορευτεί με τους άλλους φορείς ε, της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις μελέτες επαλήθευσης, θεωρούμε ότι αυτοί, αυτές θα γίνονται κατ' και από τις ε, χιλιάδες αξιολογήσεις κινδύνου που γίνονται από την ΕΦΣΑ, μόνο επτά ε, άφηναν περιθώριο για αμφισβήτηση, δηλαδή υπήρχε μία ε, ε, ε, παρέκκληση, μία μία αποδοχή από τα κράτη μέλη. Συνεπώς δεν νομίζω ότι αυτό θα χρησιμοποιείται ακτικά. Στην ουσία θα πρέπει να δίνεται επιπλέον διαβεβαίωση η ΕΦΣΑ δεν θα χρησιμοποιήσει μία θετική αξιολόγηση κινδύνων εκτός αν υπάρχει βεβαιότητα ότι χρησιμεύει. Ακόμα και όμως και σε αυτή την περίπτωση οι ε, πολίτες χρειάζονται επιπλέον διαβεβαίωση και οι φόβοι τους φόβους αυτούς θα τους ασπαστεί και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, τους φόβους των πολιτών, γιατί υπάρχει ένας οριζόντιος προβληματισμός σε όλα τα θεσμικά όργανα. Μερικοί από εσά πράσατε ε, κάποιο προβληματισμό για την πρόσβαση στα έγγραφα και την ε, επίβλεψη των ε, δεδομένων. Δεν υπάρχει τίποτα στην πρότασή μας που να υπονομεύει τις υπάρχουσες διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα. Κάνουμε το Σεπτέμβριο μία συνάντηση με την ευκαιρία το έγγραφο που κυκλοφόρησε και που προκάλεσε κάποιο προβληματισμό. Το συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη και ε, μας είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, από τις νομικές συμβουλές και νομίζω ότι πορευτήκαμε καλά. Ε, αν ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένε ε, διαστάσεις, ε, έγινε μία μνήα στο άρθρο 39 και στο 41 που θα πρέπει ενδεχομένως, θα πρέπει ενδεχομένως να παραπέψουμε, θα το κοιτάξουμε. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην εισάγουμε, ε, να μην εισαγάγουμε έναν ιό μέσα σε αυτή την πρόταση. Ενδεχομένως αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί. Ένα άλλο θέμα που ε, τέθη συχνά αφορά την ανταγωνιστικότητα για το Ε. Η Επιτροπή πραγματικά πραγματικά ε, ε, ενδιαφέρεται το θέμα της εξοικονόμησης των τροφίμων, αλλά και στην προστασία της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανία τροφίμων. Και κατά την άποψή μας δεν είναι ασύμβατα αυτά. Θα έλεγα ότι είναι απόλυτα σύμβατα για να ισχύουν το ένα το άλλο. Ε, και ένα από τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τροφίμων είναι η φήμη που έχει για ποιότητα και ασφάλεια και αυτό βεβαίως ε, σας δίνει τη δυνατότητα για πλεονάσματα στον τομέα, τον, ε, τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα και στην ασφάλεια των ε, τροφίμων. Σε ένα σεμινάριο πρόσφατα συζητήσαμε τα δεδομένα που αφορούν ε, που προκύπτουν από τα τρόφιμα. Αυτό είναι θέμα στην Ευρώπη. Η, η θάνατη αποδηλητηρίαση δεν είναι, δεν είναι πρόβλημα γιατί είναι ε, ε, είναι ασφαλή τα, τρόμα, τα τρόφιμα. Και πραγματικά όλοι, όλοι μας απασχολεί το θέμα της προστασίας. Κατά την άποψή μας η δέσμευση αυτή δεν έχει Λοιπόν από τις διατάξεις που αφορούν την διαθεσιμότητα μελετών. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά, ε, επί πραγματικά συμφωνώ. Η Επιτροπή δεσμεύεται να κοινοποιήσει μελέτες από τη στιγμή που θα έχει τους φακέλους τη διάθεση. Θα πρέπει να σας ζητήσω να συντομεύετε, γιατί πραγματικά έχουμε προς το τέλος ε, τις ε, συνεδρίες και θα πρέπει το τελευταίο λόγο βέβαια να έχει η συγκήτρια. Ε, με το σημαντικό αυτό σημείο. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι διατάξει για την προστασία των δεδομένων και ιδιαίτερα το θετικό κατάλογο επιτρέπουν στις εταιρείε να επιστρέψουν τα εμπορικά ε, συμφέροντά τους και, και στην ουσία θα καταλήξουμε με μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα βελτιώσει την αξιοπιστία όλου του συστήματος. Και αυτό βεβαίως θα έχει σαν αποτέλεσμα την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας. One minute. Ευχαριστούμε. Η συγκέντρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. τι γίνεται τώρα με αυτές τις μελέτες αντικτύπου που λείπουν. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα ήταν πολυτέλεια και μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, μα είναι απίστευτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να έχει μελέτες αντικτύπου. Αυτό συνδέεται με την καλύτερη ε, ρύθμιση και νομοθέτηση. Και ναι, θα προτιμούσα να είχα μια τροπολογία και να πέριπτα την πρόταση αυτή, γιατί δεν έχουμε μελέτη αντικτύπου. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας τα παρουσίασε έτσι ε, τόσο ωραία πριν από τις εκλογές και όλοι είναι σε διάθεση προεκλογική, οπότε θέλουν να δούνε πόσο καλά μπορούν να πουλήσουν αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό εγώ το ζήτησα. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα το δούμε και στην συνάντηση των σκιωδών πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα επίσης θυμάμαι και μια άλλη μεγάλη υπόθεση, όπου τότε η Επιτροπή στην αρχή της τελευταίας νομοθετικής ε, περίοδου δεν ολοκλήρωσε. Μπορεί να γίνει το ίδιο και αυτή τη φορά με, αυτή αυτό το θέμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε εδώ η συνεδρίαση και ευχαριστώ και τους διερμηνείς,